on at the end we, we do the. We, we, add it. We, we add your name. Don't worry. Yeah, uh, we can add still for the. In the committee we can. Yes. Okay. Okay. okay. Θα ήθελα να αρχίσουμε την συνεδρίαση, αλλά ίσως έχουμε και μια ψηφοφορία. Προσοχή. Και το Κοινοβούλιο αποφάσισε τώρα ότι πάντοτε, πάντοτε γίνεται ονομαστική ψηφοφορία στο τέλος της ψηφοφορίας, ηλεκτρονική δηλαδή, και επομένως κοιτάξτε να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Θα ήθελα πάντως όπως είπα τώρα να αρχίσω την ε, συνεδρίαση. Πρώτα λοιπόν με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως που ως συνήθως έχει διανεμηθεί ήδη πρώτη συνεδριάσεως και θα ήθελα να προτείνω δύο αλλαγές. Πάντως πιο συγκεκριμένα στα διάφορα θα ακούσαμε την κυρία Σπινέλη η οποία εξεπροσώπησε την Επιτροπή μας στην Ρώμη, στο Συμβούλιο Υπουργών εξωτερικών, όπως είπα στα διάφορα. Αν δεν προτείνει κανείς άλλη αλλαγή, τότε εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Θα ήθελα επίσης στο υπαριθμό 3 ανακοινώσεις της Προέδρου να σας πληροφορήσω ότι όπως αποφασίσαμε τον Ιούλιο, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές το πρωταθέν χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων για το 2015 που ακόμα δεν καταφέραμε να τα περάσουμε όλα. Πάντως κάποιες συνεδριάσεις που ήταν ε, χωρισμένες σε δύο διαφορετικές ημέρες τις βάλαμε Οκτώβριο και Νοέμβριο και τις έχουμε συνδέσει έτσι. Αυτό εγκρίθηκε πάντως. Θα δείτε το χρονοδιάγραμμα του 2015 αγωνιζόμαστε ακόμα να επιφέρουμε αλλαγές ακόμη σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, ωστόσο δεν έχουμε επιτύχει σε όλα. Για την ώρα λοιπόν αυτές είναι οι μόνες αλλαγές που έχουμε επιτύχει. Στο 4 τώρα, σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών, έχουμε τρία θέματα πιο σημαντικά για σας. Συζητήσαμε τις ακροάσεις για φέτος, Δύο συνεδριάσεις έχουμε όπου μπορούμε να διεξαγάγουμε ακροάσεις ή εργαστήρια Νοέμβριο και Δεκέμβριο γιατί για τον Οκτώβριο είναι πια πολύ αργά. Οι συντονιστές σας προτείνουν το εργαστήρι του Policy Department όπου θα συζητηθούν διάφορα θέματα σχετικά με τις μελλοντικέ μας δραστηριότητες, αυτό είναι το ένα, και άλλη ξεχωριστή ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Δίκαιο. Αυτά για φέτος. Άλλες προτάσεις θα συζητηθούν στα πλαίσια των αποφάσεων που θα λάβουμε για τις ακροάσεις που θα γίνουν του χρόνου. Συζητήσαμε επίσης τις γραπτές ερωτήσεις που θα υποβληθούν στον υποψήφιο επίτροπο ή στην υποψηφία επίτροπο και θα συνεχίσουμε τις επόμενες δύο ημέρες την επεξεργασία των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα ωστόσο να σας υπενθυμίσω ότι μπορούν να τεθούν και προφορικές ερωτήσεις. Άρα, οι γραπτές ερωτήσεις υποβάλλονται με, γενικό, με γενικότερο χαρακτήρα γραπτός, αλλά οι επιμέρους βουλευτές των πολιτικών ομάδων μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους χρόνο να θέσουν και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα είναι και πολιτικά χρωματισμένες και θα υπάρξει επαρκής χρόνος για να, απαντήσουν, να απαντήσει ο υποψήφιος επίτροπος. Θα διεξαχθεί και ιδιαίτερη συνάντηση των συντονιστών στο Στρασβούργο για να αρχίσει να γίνεται η συζήτηση για την εργασία μας, για τα ουσιαστικά θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή μας τα επόμενα έτη. Άρα θα γίνουν συζητήσεις αυτές και με τους συντονιστές και με τους πολιτικούς σας για να συζητηθούν τα μείζωνα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Το υπαριθμόν 5. Εδώ βέβαια λέει ώρα ψηφοφορίας. Αρχικά είχαμε προβλέψει ξεχωριστό θέμα για την συζήτηση του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είδαμε όμως τελικά ότι έχουμε μόνο μισή ημέρα συνεδριάσεως και έτσι το περιορίσαμε. Βεβαίω θα γίνει και συζήτηση, δεν είναι μοναχά η ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ ότι στην τελευταία μας συνεδρίαση του Ιουλίου συμφωνήσαμε εισηγητής για τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Συνταγματικών για τον προπολογισμό του 2014 να είναι η πρόεδρος της Επιτροπής για το θέμα ήταν κατεπήγον και ήδη είχε γίνει κάποια σχετική εργασία από την προηγούμενη Επιτροπή, δηλαδή είχαν εντοπιστεί τα διάφορα θέματα. Είχε στείλει και μια επιστολή ο προηγούμενος πρόεδρος της Επιτροπής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Άρα κάποια δουλειά είχε ήδη γίνει και συμφώνησα λοιπόν να το αναλάβω το έργο αυτό εγώ για λογαριασμό της Επιτροπής Συνταγματικών. Η καιρή είναι δύσκολη, δεν θα είναι βέβαια έτσι κάθε χρόνο. Αυτά, η δυσκολία αυτή είναι λόγω των εκλογών, της περίοδου των εκλογών. Έχουμε λοιπόν λίγο περιορισμένο χρόνο για την σύνταξη των γνωμοδοτήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ένα πρόσθετο πρόβλημα ένα εμπόδιο είναι ότι και το Συμβούλιο έχει καθυστερήσει την δουλειά του και μόλις το Συμβούλιο και μόλις τον Ιούλιο με συγχωρείτε, μόλις τον Ιούλιο οι μόνιμοι αντιπρόσωποι κατέληξαν στην θέση σε κοινή θέση το Συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα όπως πάντα θα τηρήσει την κοινή αυτή θέση. Έτσι εμείς αντιδρούμε στην απόφαση του Κορεπέρ που λήφθηκε τον Ιούλιο. Εδώ συνδέεται και η αίτησή μου προς εσάς, από πλευράς μου εισηγητρίας δηλαδή, εάν υπάρξουν κάποιες όχι ουσιώδεις αλλαγές, όπως ελπίζω, που θα επιφέρει το Συμβούλιο στο κείμενο των ε, μονίμων αντιπροσώπων και αν χρειαστεί από τη δική μας κάποια πλευρά κάποια τροπολογία ή κάποιες τροπολογίες για τη γνωμοδότησή μας, ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι αν δώσετε την έγκρισή σας στην πρόεδρο ως εισηγήτρια να επιφέρει τις ε, σχετικές αλλαγές στα όσα θα εγκρίνουμε σήμερα, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεδριάσει πρώτα η Επιτροπή μας. Εγώ βέβαια θα διαβουλευθώ με τους ε, συντονιστές, αν και ελπίζω να μην χρειαστεί. Θα χρειαστεί λοιπόν να λάβετε απόφαση σχετικά. Έχουμε διανύμει το σχέδιο της γνωμοδοτήσεως και τις τέσσερις τροπολογίες και έχουμε λάβει μόνο από την ομάδα ECR, τον κύριο Μέσσερ Σμιτ, τροπολογίες και για τον προπολογισμό και για την γνωμοδότηση και όλες οι πολιτικές ομάδες είχατε τη δυνατότητα να τα συζητήσετε. Στην γνωμοδότησή μου εκφράζω κυρίως την απογοήτευσή μας σχετικά με όλες τις καθυστερήσεις που δεν οφείλονται βέβαια όλες στις εκλογές, γιατί για τις εκλογές δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει κανένα. Δεύτερο, εκφράζω την άποψη ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στο έργο του Συμβουλίου, διότι στο Συμβούλιο οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με γραπτή διαδικασία. Και αυτό είναι σημαντικό βάρος για, μια τέτοια, για ένα τέτοιο σημαντικό θέμα όπως είναι ο προϋπολογισμός του 2014. Εκφράζω επίσης πάντοτε για λογαριασμό σας την απογοήτευση λόγω των περικοπών που γίνονται στα κονδύλια του τίτλου 3 ασφάλεια και ηθαγένεια που είναι δικές μας αρμοδιότητες καθώς επίσης εκφράζω την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για κάθε τι που έχει σχέση με την ενδυνάμωση, το empowerment αυτών των πολιτών και την χρηματοδοτική στήριξη κάθε ενέργειας που έχει σχέση με την συμμετοχική δημοκρατία. Εκφράζω λοιπόν την απογοήτευσή μας και σε ό,τι αφορά το χρηματοδοτικό και την ε, ποιότητα της χρηματοδότησης αυτής. Αυτά με λίγα λόγια διαλαμβάνονται στην γνωμοδότησή μου. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο και σε όσους και όσους εκ των συναδέλφων επιθυμούν να συμβάλλουν. Γιο Λάινεν. Οι συντονιστές δεν ζητούν τον λόγο, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ και για την έκθεση που μας υποβάλατε. Βέβαια, είναι μια ιστορία παθών που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Το Συμβούλιο προβαίνει σε περικοπές για την επικοινωνία με τους πολίτες, για τη συμμετοχή των πολιτών κλπ. Και το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να διορθώνουμε τις περικοπές αυτές. Να τις επαναφέρουμε δηλαδή στο επίπεδο του προηγουμένου έτους και ίσως να προβλέπουμε και ένα μικρό περιθώριο. Γνωρίζουμε όλοι βεβαίω ότι αυτά δεν αρκούν. Είδαμε και την εμπειρία των ευρωεκλογών ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ του έργου μας εδώ και των όσων γνωρίζουν οι άνθρωποι για το τι κάνουμε εδώ. Για την αίσθηση που έχουν ότι μένουν απ' έξω. Πρόκειται για ένα θλιβερό κεφάλαιο. Καμιά φορά χρειάζεται το θάρρος να κάνουμε περισσότερα πράγματα από ότι μια απλή επαναφορά, μια διόρθωση δηλαδή των περικοπών του Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε περισσότερο δυναμικό και για ενημέρωση των πολιτών και για τη στήριξη των συμμετοχής τους. Έχουμε μαζί μας τώρα ως Ευρωβουλευτή την πρώην Επίτροπο, ίσως μπορεί να πει κάτι γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι τα κονδύλια δεν αρκούν. Όλοι μας λαμβάνουμε καθημερινά αιτήσει να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες πολιτών διαμεθοριακές. Και αυτό σπάνια πετυχαίνει, διότι ο προπολογισμό που διαθέτουμε είναι στην πραγματικότητα απλά συμβολικός, δεν έχει καμία ουσιαστική αξία. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε την πρόκληση αυτή και προς την Επιτροπή, στον ψήφιο επίτροπο τέλο πάντων, για να καλύψουμε αυτά τα ζητήματα που αναφέρεται. Κάποιο άλλο σχόλιο. Παρακαλώ. Πέτερ Μάχ από το στην Ευρώπη των Ελευθεριών. Στο σημείο που αναφέρεται ότι με τη μικρή συμμετοχή στι ευρωεκλογέ ε, ένας πιθανός λόγος να είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Αλλά θα ήθελα να πω ότι στην πράξη δεν σχετίζεται με την έλλειψη ενημέρωσης ή μικρή συμμετοχή. Πιστεύω ότι η συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές εκλογές σε όλες τις χώρες μειώνεται. Δεν είναι αφορά μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο ένα και περισσότερο υπάρχει αυξημένη επιφυλακτικότητα, σκεπτικισμό. Δεν πρέπει να το φορτώνουμε αυτό στην έλλειψη ενημέρωση των πολιτών. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι η βασική αιτία της έλλειψης συμμετοχής στις ευρωεκλογέ η έλλειψη ενημέρωσης, αλλά είναι δείγμα του σκεπτικισμού που υπάρχει έναντι της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν έχουν λύσει τα προβλήματα που επηρεάζουν τους πολίτες. Δεν σύμφωνο λοιπόν με αυτό που αναφέρεται στο σημείο 6. Δηλαδή δεν είναι θέμα έλλειψης ενημέρωσης. Βεβαίω κάθε πολιτική ομάδα έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη που έχει. Άλλα σχόλια. Ε, η ψηφοφορία είναι σε 3-4 λεπτά, γι' αυτό να τελειώνουμε. Βίβιαν, συγγνώμη, δεν σε είδα, η κυρία Ρέντινγκ. επειδή ο συνάδελφός μου Γιώ Λάινεν απευθύνθηκε μέσα σε μένα ως πρώην επίτροπο. Έχω να πω το εξή. Ως επίτροπος, όταν έχετε ξαφνικά 25% λιγότερα κονδύλια, δεν μπορεί κανείς να τα αυξήσει τα κονδύλια αυτά, είναι υποχρεωμένος ή υποχρεωμένη να διαγράψει κάποια πράγματα τα οποία είναι λιγότερο αποδοτικά. 25% είναι πολλά χρήματα, έτσι. Εγώ είχα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στη δραστηριότητά μου σε ορισμένα πράγματα. Τώρα, εάν αυτό το κρίνετε ως λάθος εσεί είναι δική σα υπόθεση. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Remembrance. Εκεί εγώ τα ενίσχυσα όσο μπορούσα. Δεν περιέκοψα τίποτα, διότι θεωρώ ότι οι νεότερες γενιές πρέπει να γνωρίζουν από πού προέρχονται και ποιε είναι οι ρίζε του τη εδώ Ευρώπης που ζούμε. Στρατόπεδα συγκέντρωση και ούτω καθεξής στοιχεία δηλαδή ενημέρωσης γύρω από αυτά τα θέματα. Επίσης, δύο χρόνια πριν από τις εκλογές είχα αρχίσει τους διαλόγους με τους πολίτες. 51 συνολικά με εκατομμύρια συμμετέχοντες, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω διαδικτύου. Αυτά πρέπει να τα συζητήσετε κάποια στιγμή, γιατί ήταν πραγματική επιτυχία και πολλοί μας είπαν ότι για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ερωτήσεις και να λάβουμε απαντήσεις από πολιτικούς. Συμμετείχαν σε αυτές πολιτικοί της Ευρώπης, υπουργοί, εθνικοί, ε, πολιτικοί, άνδρες και γυναίκες, κάθε πολιτικής απόχρωσης. Εκεί είχα δώσει εγώ πολλά κονδύλια για να ξεκινήσω την πρωτοβουλία αυτή και να δω αποδίδει ή όχι. Απέδωσε τελικά. Αυτό που δεν έκανα ήταν αυτό το πασπάλισμα που λέμε, δηλαδή λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ένα ευρώ εκεί, ένα ευρώ εδώ και ούτε καθεξής. αυτά δεν έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα, τελικά απορροφούν πολλά χρήματα και δεν αποδίδουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες δράσεις και αυτές να τις προωθούμε και να τις φέρνουμε και σε πέρας και μετά να ελέγχουμε αυτή η διεξαγωγή τη συγκεκριμένη δράση τι απέδωσε. Αυτό καμιά φορά δυσμονείται, αυτό ο τελικό έλεγχο δηλαδή. Ευχαριστώ. Σχόλια, άλλα σχόλια. Ωραία, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ας κάνουμε έναν έλεγχο του κατά πόσον δουλεύουν τα μηχανάκια σας.

Υπάρχουν 24 άτομα που έχουν ψηφίσει, που θα μπορούσαν να ψηφίσουν και δεν έχουν. Πατήστε ό,τι θέλετε. Ναι, συν, πλην. Α, ξεχάσετε την κάρτα σας. Θα προσθέτουμε λοιπόν τον κύριο Ρανζέλ στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. 18 δεν ψηφίσατε. Πολλοί σοσιαλιστές. Βγάλτε ένα σοσιαλιστής την κάρτα. Έγινε εντάξει. Εσεί που δεν ψηφίσετε υποθέτετε ότι λειτουργεί το μηχάνημά σα χωρί πρόβλημα. Εντάξει. Δεν ξέρω πού κάθονται οι συντονιστέ, συγγνώμη γι' αυτό. Θα πάμε αργά αργά αυτή τη φορά. 69.00 υπέρ. Τροπολογία 69.00 υπέρ. Κατά. Κατά. Εγκρίνεται. 6904. 6904. Υπέρ. Κατά. Ας κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. 6904. Άρχεται η ψηφοφορία. Συν για όσους είναι υπέρ, μείον για όσους είναι κατά. Δεν ψηφίσατε όλοι, αλλά πρέπει να λήξει ψηφοφορία. 11 υπέρ 69-01 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69-03 υπέρ Κατά. σεφ Εγκρίνεται. Τώρα. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δύο. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της δεύτερης τροπολογίας. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά νομίζω. Και για τα δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα τη δεύτερη τροπολογίας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Δεύτερο τμήμα τη δεύτερη τροπολογίας. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται με διαφορά. Το δεύτερο τμήμα. Τρία. Τρίτη τροπολογία, υπάρχει και προφορική τροπολογία, εάν κατάλαβα καλά, από και δημοκράτες. Παραδοσιακά δεν παρουσιάζονται στην Επιτροπή οι προφορικέ τροπολογίες. Υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται στην προφορική τροπολογία. Όχι, οπότε ψηφίζουμε την τρίτη τροπολογία όπως τροποποιήθηκε προφορικός. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, Νομίζω γκρίνεται. Δεν ζητάει κανεί έλεγχο. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Νομίζω γκρίθηκε. Αλλά ας ελέγξουμε για την τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. Και μετά 10. Πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω να κάνουμε έλεγχο. Πρώτο τμήμα της 10 τροπολογίας. Πέρας. Απορρίπτω. Όχι. Πολ είσαι υπέρ. Ωραία λοιπόν. 9 προς 10. Ο Πάολο Ραζέλ έσωσε την τροπολογία. Το πρώτο τμήμα τουλάχιστον. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική. Α, είναι απλώς νομοδότηση. Ωραία. Ηλεκτρονικός λοιπόν ψηφίζουμε. Ναι, μόνο για τις νομοθετικές έχετε δίκιο. Πέρασε. Εγκρίνεται. 17 προς 3. Εγκρίνεται. Περνάμε στα διάφορα. Στο σημείο 6 σας ενημέρωσα για τη συζήτηση που είχαμε Είχαμε μετρήσει έναν επιπλέον γιατί ο κύριος Ρανζέλ δεν είχε κάρτα προχωρίας μαζί του. Εντάξει. Περνάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Διάφορα. Εδώ θα ήθελα κυρία Σπινέλη που συμμετείχε εκ μέρους μας στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στη Ρώμη α, τέλη Αυγούστου θα ήθελα να μας ενημερώσει για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου εκεί. Μπάρμπαρα. Στο Μιλάνο, με συγχωρείτε. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε που δεν θα εκφραστώ στα αγγλικά. Θα, προσπαθώ, θα προσπα... προτιμούσα να είμαι ελεύθερη στην έκφρασή μου. Πριν ανακεφαλαίωσω λοιπόν τα συμπεράσματα του επισήμου Συμβουλίου στο Μιλάνο και τις δικέ μου τοποθετήσει εκ μέρους του Κοινοβουλίου, μια εισαγωγή, εισαγωγική παρατήρηση. Επειδή δεν είχα λάβει συγκεκριμένη εντολή από αυτήν την ε, επιτροπή, θύμισα ποια είναι η βασική της αποστολή, μεγαλύτερη διαφάνεια, συμμετοχή, συμμετοχή των πολιτών, ε, να προβλέψουμε τι θα μπορούσε να γίνει εφόσον οι συνθήκες παραμένουν ως έχουν ή εφόσον υπάρχει τροποποίηση. Αλλά μετά σε προσωπικό επίπεδο έκανα και κάποια παρέμβαση μιλώντας για τη βαθιά κρίση την οποία διανύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη λειτουργία της και κυρίως το μήνυμα που μας έχουν αποστείλει οι πολίτες και μας το απέστειλαν πολύ ξεκάθαρα στις 25 Μαΐου. Αυτή λοιπόν την παρουσίαση θα ήθελα να τη διαιρέσω σε δύο τμήματα σε μια πρώτη φάση το τι συζήτησαν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που βρίσκονταν εκεί και έπειτα να αναφέρω σε δεύτερη φάση τι έθιξα εγώ κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πρώτον, η γενική εντύπωση που είχα είναι ότι οι υπουργοί ανησυχούσαν ε, για την ε, κρίση εμπιστοσύνης που διαφάνηκε μέσα από τις τελευταίες εκλογές. Όμως δεν έχουν και συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν απλώς μια συγκεχημένη διάθεση να υπάρξει καλύτερο συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Επιθυμούν οι πολίτες να έρθουν πάλι κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά δεν αναγνωρίζουν ότι τα ίδια τα θεσμικά όργανα καλούνται αυτά να πλησιάσουν περισσότερο τους πολίτες. Στο κέντρο της προσοχής ε, των Υπουργών ένα σημείο αναφοράς το οποίο κανείς δεν παρέβλεψε είναι η στατηγική ατζέντα που έχει εκπονήσει ο Φαναρομπόε και ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούνιο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η ατζέντα αυτή, ο κατάλογος που το ε, ήταν ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι ε, επανειλημμένως. Ο κ. Γκότζη πολλές φορές τη χαρακτήρισε βίβλο μας, το Ευαγγέλιό μας. Ε, η δική μου θέση είναι ότι μπορεί να γίνει ενός είδους ε, που μας υποχρεώνει σε συγκεκριμένες κινήσεις ε, το έγγραφο αυτό σε κοινοτικέ δράσεις και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ε, λογοτεχνική παρέκβαση, διότι στον άνθρωπο χωρίς ιδιότητες του Μούζιλ η συγκεκριμένη ε, κυριαρχία της Αυστρογγρικής Αυτοκρατορίας κλονίζεται διότι χρειάζεται μια σημαντική παράλληλη δράση πολύ συγκεκριμένη που όμως δυστυχώς δεν έχει ουσία και τελικά δεν παρεμποδίζει και την ε, ε, κατάρρευση της ε, Αυστρογκρικής Αυτοκατορίας καθώς και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η στατηγική ατζέντα του Φαρόμποι και το Συμβούλιο του Μιλάνου μου θύμισαν λίγο αυτήν την ταυτόχρονη προσπάθεια. Δεν λείπει βέβαια η συνέστηση ότι κάτι θα πρέπει να γίνει, διότι είναι πολλά τα συμβούλια υπουργών σε τομεακό επίπεδο που δεν επικεντρώνονται αρκετά στον κεντρικό ρόλο που έχει τελικά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Όπως ε, πολλές φορές συμβαίνει, ε, η μέθοδος που ακολουθείται τελικά οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Κατακαιρματισμός των ε, συμβουλίων, η ανάδειξη της διακυβερνητικής μεθόδου, η δημιουργία νέων επιτροπών και εδώ η πρόταση του Υφυπουργού Γκότζη να δημιουργηθεί μια ομάδα που να, οκαλείται να φίλη της Προεδρίας. Θα είναι μια πολλωστή προσπάθεια δημιουργίας επιτροπής όπου δεν θα ασκείται κανένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, ούτε ευρωπαϊκός ούτε εθνικός. Και είναι πολλές οι αντιπροσωπείες, όχι όλες βέβαια, οι οποίες έχουν ζητήσει ρητός το Κοινοβούλιο να μη συμμετάσχει σε αυτή την ομάδα μία ε, ενδιαφέρουσα παρατήρηση για την πρόταση αυτή ήταν αυτή του Πορτογάλου Υφυπουργού για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ότι το Συμβούλιο διακινδυνεύει να μην λειτουργήσει εφόσον δεν θα, Σωστά, εφόσον δεν θα υπάρχει ένα υπεύθυνο φορέας για να συντονίζει τα διαφορετικά σημεία λειτουργίας του. Το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, για παράδειγμα, συνολικά, αν δεν υπήρχε ολομέλεια και βασιζόταν μόνο στι επιτροπέ. Περνάω τώρα στι δικέ μου τοποθετήσει. Στην εισαγωγική μου παρατήρηση ζήτησα η στατηγική ατζέντα να μην θεωρείται ω ε, ε, ένα αυτό αλλά να αποφύγουμε το να γίνει ενός είδους υποχρεωτική πορεία, ρουλομαδίας δηλαδή. Και βλέποντας το τι συζητήθηκε και το Μάρτιο στο Συμβούλιο, βλέπουμε ότι ε, το έγγραφο αυτό διέπεται από το πνεύμα του εγγράφου του 2012, όπως είχε εγκριθεί, με τέσσερις ε, βασικές ε, προτεραιότητες και η, τα στοιχεία της κρίσης ε, του ευρώ, δηλαδή οι ανισότητες και ανομοιότητες μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με το ευρώ, ε, είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη σε πολιτικό επίπεδο για την Ευρωζώνη. Η βασική μου λοιπόν επικριτική παρατήρηση ήταν ότι ε, ήταν τιμωρητική η ψήφος των ε, ψηφοφόρων στις 25 Μαΐου προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αλλά ακόμη συνεχίζει να υποτιμάται η κίνησή τους. Κάποιοι που ε, λέγαν ότι ε, ουσιαστικά απογοητεύτηκαν από το πνεύμα της στρατηγικής ατζέντα, τώρα πια αποκαλούνται ε, λαϊκιστές οι εξτρεμιστές, ενώ πολλές φορές είναι απλώς επικριτές της Ευρώπης, είναι απλώς εχθρικοί προς την Ευρώπη. Κατήγγειλα κάποιες αντιφάσεις επίσης στα λόγια που ακούμε πολλές φορές στα άτυπα συμβούλια, διότι ενώ ε, κάποιες κυβερνήσεις όπως η Γαλλία αρχίζουν να περνάνε σε μια κρίση, ενώ οι υπουργοί οικονομικών που αυτή τη στιγμή ο κύριος Παντοάν, ο, που προεδρεύει στο ΕΚΟΦΗΝ, όλοι παραδέχονται ότι ε, σφάλαμε στις προβλέψεις για την ε, ανάπτυξη και οι διεθνείς οργανισμοί και οι κυβερνήσεις και ούτω καθεξής, όλες συνεχίζουν να δείχνουν συγκατάβαση και να χαίρονται με τα αποτελέσματα που έγινε για τη μείωση του κρατικού χρέους στα διαφορα κρατημέλη και με τις πολιτικές λιτότητας. Έτσι λοιπόν εξέφρασα την ελπίδα ε, ο κύριος Γιούνκερ να προβλέψει ένα κοινό πρόγραμμα επενδύσεων στην πραγματική οικονομία με 300 δις ευρώ ετησίως. Κάτι στο οποίο θα πρέπει να δεσμευτούν όλες οι κυβερνήσεις. Προσωπικώς βεβαίως θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθούν τα απαραίτητα μέσα για κάτι τέτοιο. Ε, επίσης επέμεινα σε ορισμένα σημεία όπως την διαφάνεια και τη συμμετοχή. Ε, το κοινοβούλιο μας δεν μπόρεσε να ασκήσει έλεγχο ούτε στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ούτε στην ε, Τραπεζική Ένωση, ούτε θα μπορέσει να το κάνει αυτό στο επίπεδο των φίλων της Προεδρίας, ούτε στην ε, διατλαντική διαπραγμάτευση για το εμπόριο, δηλαδή το TTIP, και ε, παρόλο που η Ιταλική Προεδρία ζήτησε σωστά ε, να ε, τροποποιηθεί η διαβηματευτική εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συστηματικά επίσης παραβλέπεται το άρθρο 11 της Συνθήκης της Λισαβόνας, το οποίο υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα να τηρούν διαρκή ανοιχτό και συστηματικό διάλογο με τις ενώσεις εκπροσώπησης των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό μας θύμισε προλίγου μόλις ο συνάδελφος Γιώ Λάινεν. Και ενώ η ατζέντα αυτή υποσχόταν ε, κάποιες αλλαγές, όπως την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, του περιορισμού των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, αυτά δεν αναφέρθηκαν πουθενά στα έγγραφα της Συνόδου του Μιλάνου. Η ατζέντα αυτή καλούσε την Ένωση να ενισχύσει τις πολιτικές του ασύλου, ενώ την παραμονή της ε, συνεδρίασης στο Μιλάνο η επιχείρηση Search and Rescue αναζήτησης και διάσωσης των μεταναστών στο Mare Nostrum δεν ξέρουμε κατά πόσον μπόρεσε να έλθει εις πέρας και με τι πόρους. Ε, μόνο η πολιτική απόθεσης μπόρεσαν να στηριχθούν. Στην συζήτηση για την αλλαγή στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνω, σημείωσα μάλλον ότι όλοι ε, λυπούνται για τον καταγραμματισμό της λειτουργίας του ανατομέα δράσης αλλά αναγκάστηκα και εγώ να θυμίσω ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει μακρά ιστορία και πείρα σε αυτόν τον τομέα. Ε, ήδη δύο φορές προτάθηκε ως λύση να ενοποιηθούν τα τομεακά συμβούλια και να υπάρχει ένα ενιαίο νομοθετικού χαρακτήρα συμβούλιο. Έτσι θα καταλήγαμε, ε, όπως μάλλον ε, στην είδη στο Κοινοβουλίο το 1974, στο σχέδιο συνθήκης που είχε οδηγήσει στη δημιουργία αυτή, τέτοια πρόταση που είχε ξαναυποβληθεί το 2003 για σύνταγμα από το 2003 τελικά παραγωνίστηκε πλήρως από τη διακυβερνητική διάσκεψη. Θύμιζα, ε, θύμισα και πάλι ως προς την ε, κακή λειτουργία των θεσμικών οργάνων ότι όπως τη συζήτηση στο Μιλάνο μεταξύ των Υπουργών έλειψε η αναφορά στον Επίτροπο που θα είναι επιφορτισμένος με θέματα μετανάστευσης το ίδιο συνέβη και τώρα και το συζητάμε εδώ και εβδομάδες χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση να γίνει κάτι γι' αυτό. Κάποιοι υπουργοί μάλιστα μιλήσαν για εξωτερική πολιτική και τους διάφορους πολέμους που μας αφορούν. Εδώ λοιπόν θύμισα ότι η Ένωση δεν έχει αρκετές ιδέες σε αυτόν τον τομέα, ιδίως στο τι θα κάνει στις σχέσεις της με, της με τη Ρωσία. Ε, ολοκληρώνοντας, ε, και εδώ διαπίστωσα ότι υπήρξε αρκετή αυτοκανοποίηση ε, στο επίπεδο του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων και όπως και στην περίπτωση της συζήτηση για τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι περισσότεροι θέλουν να παραμείνουν στο πεδίο της συνθήκης αυτής, αποφεύγοντας τις αλλαγές. Μόνον λίγοι είναι αυτοί που αναφέρονται σε αλλαγές, αλλά πολύ μακροπρόθεσμα. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, για να δώσω ένα παράδειγμα, σημειώθηκε η ταχύτητα με την οποία η Ένωση ενέκρινε ε, προτάσεις κυρώσεων και επιβολή τιμωριών για την Μόσχα. Αυτήν την ικανοποίηση της Ένωσης δεν τη συμμερίζομαι. Οι κυρώσεις δεν είναι ανάλογες μιας συγκεκριμένης και διαρθρωμένης πολιτικής προς τη Ρωσία ή την Ουκρανία. Η ε, Frontex, η ομάδα κρούσης για τη Μεσόγειο ε, οι, οι κινήσεις των κρατών μελών εδώ και χρόνια μεμονωμένα δεν δείχνουν να υπάρχει καμία συντονισμένη πολιτική ούτε προς τα αραβικά κράτη, ούτε προς τη Λιβύη, ούτε να υπάρχει διάθεση να ε, αγκληφθεί μέρημνα για τον πόλεμο στη λόριδα της Γάζας μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Ευχαριστούμε κύριε Σπινέλη. Θέλει κάποιος να κάνει σχόλια ή να θέσει ερωτήσεις. Να σας πω το Συμβούλιο Γενικών Προθέσεων προφανώς προσπαθεί να ανακτήσει την θέση του μέσα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ε, δημιούργησαν αυτή την ομάδα των φίλων της Προεδρίας για να εντοπίσουν μέχρι το τέλος του έτους από την κατάλαβα πιθανές αλλαγές μέσα στη συνθήκη και δεν θέλουν άλλα όργανα, δεν ξέρω για την Επιτροπή, σίγουρα πάντως δεν θέλουν το Κοινοβούλιο να εμπλακεί, Θα ήταν να ξέρουμε τα αποτελέσματα ωστόσο, τον αποτελεσμα, να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της, των εργασιών της ομάδας αυτής για τις πιθανές αλλαγές συνθήκες θα μπορούσαμε να έχουμε μία σύνδεση με την Προεδρία για το σκοπό αυτό. εν ώψη των μεταρρυθμίσεων που έχει στην μέση διαταξή το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Εμείς είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε το πώς οι σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και ημών και του νέου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξελίσσονται. Ήταν λοιπόν σημαντική η συνάντηση αυτή του Συμβουλίου. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Παύλο Ραντζέλ, που αυτός έχει επίσης ένα θέμα. Κάτι... Μια παρατήρηση μόνο. Διότι χρησιμοποιούμε αυτό το γερμανικό οργανωζατσιόν θέμα οργάνωσης. Δεν νομίζω ότι το σχέδιο χρονοδιαγράμματος είναι καλό. Θα ήθελα να το πω αυτό. Πρώτον, το σύστημα που έχουμε, που είχαμε παλιά, ένα απόγευμα ένα πρωί ήταν καλύτερο από μια συνάντηση πρωί-απόγευμα που είναι πιο απαιτητικό. Και μερικέ φορές έχουμε και κάποια πλεονεκτήματα να περνάμε μια νύχτα μεταξύ των δύο συναντήσεων να σκεφτούμε πέντε πράγματα. Επίση, το άλλο θέμα είναι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες μέρες το να πηγαίνουμε από τρίτε, δευτέρε, τρίτη, δηλαδή από δευτέρα μέχρι πέμπτη χωρίς να έχουμε συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι ε, καλό για, για μας αλλά και για το κοινό. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη μέρα συνάντησης. Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε έκτακτες συναντήσεις, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο να λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τρίτη, Τετάρτη, μόνο Τετάρτη. Κατά κανόνα. Όταν πηδάς από μέρα σε μέρα, δεν είναι πολύ άνετο. Και βεβαίω. και η εικόνα της Επιτροπής μας δεν προβάλλεται καλά διότι δείχνουμε ότι κάνουμε ό,τι μας βολεύει και όχι σε συγκεκριμένες μέρες. Όπως έχουμε εβδομάδες, εβδομάδα επιτροπών, εβδομάδα ομάδων, οι συναντήσεις των ομάδων είναι την ίδια μέρα, οι συναντήσεις των προεδρίων των ομάδων την ίδια μέρα και αυτό μας επιτρέπει να προβλέπουμε τι κάνουμε. I'm not saying that we should change this. For me... Δεν λέω να αλλάξουμε τα και καλά, αλλά δεν είναι πολύ πρακτικό. Τον ένα μήνα είναι πέμπτη, την άλλη είναι τρίτη και τα ταξίδια μας είναι προβληματικό. Έτσι το λέω. Σας είπα ότι εγώ δεν εμπλέκομαι, είναι οργανωτικό θέμα και οι συντονιστέ φαντάζομαι, αλλά ω μέλο τη επιτροπή, θέλω να το πω ρε παιδί μου. Ευχαριστούμε. Ο κ. Σέπφλιν. Uh, Σε συνέχεια αυτού που είπε ο κ. Ζανζέλ Έκαναν προσπάθεια οι υπηρεσίε να βρουν κάποιε μέρε, αλλά έχω κάποια προβλήματα για το να συναντιόμαστε πέμπτη απόγευμα. Η παρουσία θα είναι πολύ αδύνατη. Και αυτό δεν είναι καλό για τη φήμη τη Επιτροπή. Υπάρχει τρόπο να πιέσουμε ούτως ώστε να μην είμαστε πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα πάντως είναι κάτι που θα είμαστε τρει και κούκος. Σχόλια. Έγινε η συζήτηση και τον Ιούλιο. Έκανε ό,τι μπορούσε η Επιτροπή. Ξέρουμε ότι οι πέμπτες είναι πολύ κακές. Αν θέλετε να μπορεί, μόνο πέμπτες μας δώσανε. Αν θέλετε μπορεί να ε, Πάμε και Παρασκευές. Ξέρετε ότι η επιτροπή αυτή έγινε ουδέτερη αργά τον Ιούνιο, οπότε όλοι είχαν άλλες δεσμεύσει. Υπήρχαν δηλαδή προβλήματα με όλες τις επιτροπέ συνέχεια. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι η γραμματεία προσπαθεί να καλύψει και τα θέματα με τη διοίκηση είμαστε ικανοποιημένοι με πολλά θέματα. Ζήτησε από τον Ζωζέ να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Οι πιθανότητες πάντως είναι, το ξαναδεί, υπάρχουν πάντως πολλά θέματα και δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι. Τι είναι θέματα όχι μόνο συμμετοχή σε άλλες επιτροπές αλλά και τα σλότ, ε, Έχουμε να παλέψουμε και με άλλες επιτροπές. Αν η πολιτική ηγεσία σας μπορεί να κάνει οτιδήποτε για να επηρεάσει τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να αντιμετωπίσει την Επιτροπή με καλύτερο τρόπο, κάντε το. Δεν ξέρω όμως τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε κάνει μάχες πάντως για το θέμα αυτό. Ούτε οι Δευτέρες απόγευμα είναι εύκολες για πολλούς από εσά. Όπως βλέπετε οι περισσότερες συναντήσεις είναι ακόμα πέμπτες. Αυτό απαιτεί από εσά να μείνετε πέμπτες στο κοινοβούλιο. Ξέρω τι γίνεται τις πέμπτες. Να το προσπαθήσουμε, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ οτιδήποτε. Ευχαριστώ πάντως. τα συμμερίζομαι, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, αλλά αυτή είναι η ζωή. Αν νομίζετε ότι μπορούμε να, ότι μπορείτε να βοηθήσετε μέσω των πολιτικών σας ε, γνωριμιών να δώσετε καλύτερες μέρες για τις συναντήσεις της Επιτροπής, κάντε το. Αλλά σας λέω, πολύ λίγες περιπτώσεις, πολύ λίγες πιθανότητες, συγγνώμη. Σχόλια, άρα ολοκληρώνουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και την κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Θα ξανασυνεδριθούμε στο Στρασβούργο. Τέλος συνεδρίασης.